Ξεκινάμε πάλι. Θα ακούσουμε τον Ζεράρ Ντεπρέ για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης κατάθεσης της κατάθεσης αίτησης για διεθνή προστασία από τρίτη χώρα ή από απάτριδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη, λαμβάνοντας υπόψη το ότι η έκθεση αυτή, οι δύο εκθέσεις συνδέονται, είναι μια ευαίσθητη έκθεση. Θα ήθελα να δώσω την τύχη σε κάποιους συναδέλφους να έρθουν εδώ και να πάρουν το λόγο, αν υπάρχουν. Κοιτάξτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το Eurodac, το οποίο είναι λιγότερο ευαίσθητο. Καλώς, πρόκειται λοιπόν για τη δεύτερη έκθεση. Να σας θυμίσω εδώ, να θυμίσω τα μέλη. Τι είναι το Eurodac, γιατί κάποιοι ίσως να μην το γνωρίζουν. Είναι ένα συγκεντρωτικό, αν θέλετε, ηλεκτρονικό σύστημα που συγκεντρώνει τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν καταθέσει αυτοί που έχουν ζητήσει άσυλο, αυτοί που έχουν περάσει τα σύνορα παράνομα, αυτό υπήρχε σαν σύστημα έτσι και αλλιώ. και η νέα μεταρρύθμιση προβλέπει ότι θα ισχύσει και για αυτούς οι οποίοι είναι ε, σε, ε, ε, είναι σε μια χώρα παρανόμως και έχουν εντοπιστεί από τις αρχές καταστολής στο εσωτερικό των κρατών μελών. Όχι μόνο λοιπόν αυτοί που περνούν τα σύνορα, αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Διεύρυνση δηλαδή της εμβέλειας, σχετικά τώρα με τις αρμοδιότητες της δικές σας. Το συνολικό κόστος είναι λογικό 30 εκατομμύρια ευρώ σε τέσσερα χρόνια. Να κάνω όμως κάποια σχόλια για τις τροπολογίες, γιατί νομίζω ότι το ποσό αυτό τεκμηριώνεται εφόσον έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές ε, στον κανονισμό ο οποίος ε, ισχύει και που οι αλλαγές αυτές έχουν και δημοσιονομικές επιπτώσεις. Τον προτείνω τον καθορισμό της συμβατότητας ανάμεσα στον αριθμό των δακτυλικών αποτυπωμάτων από εδώ και πέρα με το σύστημα το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία εισόδου και εξόδου στις προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για το σύστημα εισόδου-εξόδου θα παίρνουμε τέσσερα αποτυπώματα και ένα αποτύπωμα προσώπου. Στο Eurodac όπως προτείνεται στη φάση αυτή θα παίρνουμε 10 δακτυλικά και ε, ένα αποτύπωμα προσώπου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε σε τέσσερα και όχι σε 10. Οπότε όταν μιλάμε για δακτυλικά αποτυπώματα θα ήθελα παρακαλώ να μιλάμε για τέσσερα. Αυτό ισχύει για τους πενταδάκτυλους λέει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, ναι, ακόμα και ένα χέρι να έχετε, λέει ο κύριος συγητής. Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με ένα στόχο εναρμόνισης και όπως σας είπα, Κάτι το οποίο δεν είναι σαφές αν θέλετε, ξεκάθαρο στην παρούσα αυτή πρόταση. Θα πρέπει να υπάρξει διαλειτουργικότητα και αυτόματη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο σύστημα εισόδου-εξόδου, το οποίο καλύπτεται από άλλον κανονισμό, και το σύστημα Eurodac. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για την έκθεση αυτή. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες, όχι σημαντικές. Η διαλειτουργικότητα ίσως να έχει ένα επιπλέον κόστος, αλλά αυτό έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Αν έχετε ένα σύστημα πληροφορικής το οποίο δεν είναι διαλειτουργικό, τότε τι νόημα έχει. Αυτά. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Δεν ξέρω, κάποιος συνάδελφο θέλει το λόγο, η κυρία Σούλινα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα σας συγγνώμη γιατί δεν ε, ζήτησα το λόγο για το πρώτο κομμάτι. Και το αλλάξατε. Α, αλλάξατε μάλλον τη σειρά, οπότε δεν έχω να πω κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος, παρακαλώ, κύριο Τινανού. Πρόεδρε, όντω ω ότι για την ομάδα μου, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά που έκανα και για την πρόταση γνωμοδότηση. Ε, και συμφωνώ με πολλέ από τι διαπιστώσει του. Το σύστημα του Δουβλίνου, με το οποίο συνδέεται το Eurodact, έχει περάσει πριν από πάρα πολλά χρόνια και έχει δείξει εξ αρχής ότι είναι δυσλειτουργικό. Δεν ήταν η επιθυμητή η επίδρασή του και σε ό,τι αφορά τους ε, μετανάστες, τους ετούντε άσυλο, επιτρέπει ουσιαστικά την επιλογή ε, το που υποβολής αίτησης ασύλου. Και το σύστημα παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι ενισχύ. η πρόταση της ε, Επιτροπής του 4 Μαΐου 2016 που έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό ρεύμα το 2015 αναφέρεται στο κανονισμό του Δουβλίνου και του Eurodac και μια πρόταση για την δημιουργία υπηρεσίας ευρωπαϊκής για το άσυλο. Θεωρώ ότι θα έχει καταρχάς το πλανέκτημα της αλλαγής και της μεταρρύθμισης προκειμένου το σύστημα να κατασταθεί πιο λειτουργικό και πιο πρακτικό. Θα ήθελα, όπως είπε και ο συγκεκριτής, να τονίσω ότι ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλάω και όχι ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Δικαιωμάτων. Άρα ουσιαστικά η δουλειά μας έχει να κάνει με την εξέταση των δημοσιονομικών επιπτώσεων και όπως είπε ο εισηγητής δεν υπάρχουν ουσιαστικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά την τετραετία αυτή περίοδο του τουλεχθέντος. Τίφονται και θέματα περιεχομένου πέρα από τα θέματα τα δημοσιονομικά. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι σήμερα υποστηρίζω την πρόθεση να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψε, ε, δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων σεβόμενοι και την αρχή του αλληλοσεβασμού και την πρόταση να μην δίδεται ε, προτού δοθούν αυτέ οι πληροφορίε στην Eurodac. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν συμφωνούμε από την ομάδα μου με την πρότασή του να συμπεριληφθεί στη βάση του Eurodac μια διαδικασία επανεκατάσταση σε ό,τι αφορά του των χωρών. Γιατί αυτό εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση και το Eurodac θα πρέπει να σεβαστεί τη συνομολογία αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να υπάρχει εντελειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την ε, υποδοχή των ε, ετούντων άσυλων και να ε, διευκρινίσουμε ότι η Eurodac δεν, δεν υποκαθιστά τις εθνικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων και τη λήψη δεκτυλικών αποτυπωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν κάποια στοιχεία προληπτικά, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά ισχύουν για όλου του μετανάστε, η όλου αυτού που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει η Μόνικα Χόλμαϊρ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ακριβή και πολύ αξιόλογη η δουλειά που έχει κάνει στο θέμα του Eurodact. Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να κινηθούμε προ τα εμπρό, δεν έχουμε άλλη επιλογή και από δημοσιονομικής πλευράς. Γιατί έχουμε διπλή εργασία σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχει μια τελειτουργικότητα με την οποία δεν θεωρώ ότι εξαντλούμε το δυναμικό που έχουμε και κατά τρίτον ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο και φυσικά ξεκινώντας από την αρχή ότι δεν είναι όλοι τρομοκράτες και για όλους τους Γάλλους και Γερμανούς επικούς έχουμε βιομετρικά διαβατηρία. Γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τους ε, μετανάστες. Χρειαζόμαστε βιομετρικά στοιχεία. Τα χρειαζόμαστε και για ποινικού λόγους. Η κατάσταση στη Γερμανία έχει ως εξή ε, στην παρούσα φάση. Όποιος έχει επιχειρήσει να εκτελέσει επίθεση είτε είναι μετανάστες είτε πρόσφυγας, ε, ήταν μάλλον είτε μετανάστες είτε πρόσφυγας και μερικές ε, περιπτώσεις με βοήθεια Γερμανών πολιτών. Δεν θέλουμε φυσικά να καταδικάσουμε ολόκληρες ομάδες κατά Αλλά Όταν μιλάμε για το φόρους, για παράδειγμα, κάνουμε έλεγχο διαρκώς. Γιατί μιλάμε για χρήματα και τα χρήματα θέλουμε να τα ανακτήσουμε σε περίπτωση που είναι χαμένα έσοδα. Αλλά όταν Μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ. Διστάζουμε σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σφαίρα των δεδομένων. Θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη η προσέγγιση. Το λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες από δημοσιονομική άποψη, Είναι και αναλογική και θεωρώ ότι ανταποκρίνεται και στις ανάγκες τις σημερινές. Και μας επιτρέπει να εργαστούμε αποτελεσματικά. Και πραγματικά στο μεγαλύτερο τμήμα δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Το θέμα με τα τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα να το συζητήσουμε για να δούμε κατά πόσον αρκούν σε περίπτωση που παρουσιαστεί κίνδυνος και κατά πόσον έχει νόημα. Δεν μπορώ να αποφανθώ στην παρούσα φάση. Θα έπρεπε να το συζητήσουμε και με τις αρμόδιες αρχές, όπως είναι η Frontex, οι συνοριοφύλακες. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Και από αυτό θα εξαρτηθεί και το τι θα αποφασίσουμε. Και πιστεύω ότι το σύστημα Eurodac και για λόγους αποτελεσματικότητας θα πρέπει να συντονιστεί καλύτερα με το ΣΥΣ για να διαπιστώνουμε κατά πόσον κάποιος έχει διαπράξει κάποια επίθεση. Και όταν ελέγχεται ένα φορολογούμενο για το κατά πόσον έχει πληρώσει καλά του φόρου του και περνάει από επιθεώρηση και από έλεγχο, δεν σημαίνει ότι τον υποπτευόμαστε και τον κατηγορούμε για φοροδιαφυγή. Όχι. Απλά ξέρουμε ότι πάντα, ακόμα και από τους κανονικά φορολαγούμενους, προκύπτει σφάλμα ή απάτη. Και φυσικά ότι ο πιο πολλής κόσμος πληρώνει κανονικά τους φόρους τους. Το ίδιο ισχύει και για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες. Θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό για κάποιο άνθρωπο Μπορεί ναι, μεν να διώκεται, μπορεί να έχει φύγει από την πατρίδα τώρα, παρόλα αυτά και μεταξύ αυτών, όπω μεταξύ των φορολογούμενων υπάρχουν και αυτοί που δεν πρέπει να πάτε, μεταξύ αυτών των ανθρώπων υπάρχουν και κάποιοι που είναι ύποπτοι. Μιλάμε λοιπόν για τα θέματα καταχώρηση και διαλειτουργικότητα με άλλε βάσει δεδομένων. Και την ανταγωνισμό με το Schengen Border Code, σύμφωνα με τον οποίο οποιοδήποτε περνάει τα σύνορα, θα πρέπει να ελέγχεται για το κατά πόσον έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Είτε είναι Ευρωπαίος πολίτης, είτε είναι κάτοχος βίζα, είτε είναι πρόσφυγας, είτε είναι κάποιος που δικαιούται να ταξιδέψει χωρίς βίζα. Όλοι θα πρέπει να περνούν από έλεγχο για το κατά πόσον διώκονται. Αυτό είναι δυνατόν με τους σύγχρονους ελέγχους. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε μία πλήρη επισκόπηση της κατάστασης χωρίς να απευθύνουμε κατηγορίες και υποψίας. Και αυτό με τα τέσσερα τελικά αποτυπώματα θα ήθελα να το συζητήσουμε λοιπόν. Και νομίζω ότι όντω οι προσεγγίσεις των, ε, του και σε ό,τι αφορά τις 15 ημέρες για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Να δούμε κατά πόσον ε, εθελοντικά μετακινείται ή κατά πόσο θα πρέπει να καταχωριστεί στο γυροντάκι γιατί ενδεχομένω να είναι τον άσυλο ο υποψήφιο. Ή υπάρχουν άλλοι λόγοι και αιτίε. Θεωρώ ότι 15 ημέρε είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Και για ω περιορισμό και σε περίπτωση που έχει ασκηθεί, έχει γίνει απόπειρα χτύπηματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκόλμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συναδέλφο Ντεπρέ για το σχέδιο έκθεσης αυτό. Γιατί όχι μόνο γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πιστεύω ότι όντω αποτελεί ένα σημαντικό θα λίθο για αυτό που ανέφερα σήμερα το πρωί. Για μια στρατηγική για την συνολική μεταναστευτική κρίση. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε ε, αξιόπιστοι, γιατί δεν αντιλαμβάνεται ο πολίτη πλέον καθόλου πώ είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε και να δρούμε με διαφορετικό τρόπο. Όλοι ξέρουμε αναφορές και περιστατικά σε ό,τι αφορά όχι μόνο την τρομοκρατία, αλλά και για δημόσιες υπηρεσίες, όπου ήταν πραγματικά ανεπαρκής ο έλεγχος και τα όσα έγιναν. Και το θέμα δεν είναι ότι είμαστε, υποπτευόμαστε τους πάντες και τα πάντα. Το θέμα είναι ότι το μεγαλύτερο τμήμα των μεταναστών δεν θα πρέπει να το θεωρούμε ύποπτο, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να εντοπίσουμε και τα μαύρα πρόβατα. Μα για, τον τρο... για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει καταχώρηση και θα πρέπει να συμβαίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν. Γιατί όλοι όσοι ταξιδεύουμε ξέρουμε ότι όταν πάει κανείς στη ΣΥΠΑ είναι απαραίτητο στο αεροδρόμιο να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Όλοι τα ζούμε, όλοι τα δεχόμαστε αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να τα αποδεχτούμε αυτά και να τα πετύχουμε και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πήραν το λόγο όλοι και να δώσουμε τώρα το λόγο στο συντάκτη της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέρφους που μπήκαν στον κόπο να δείξουν ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και να κάνουν παρατηρήσεις. Ε, για να απαντήσω στις παρατηρήσεις τους θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα ώστε να είναι σαφή κυρίως ε, για τα όσα είπε ο κύριος Δενανό. Το Eurodac δεν είναι ε, εργαλείο ασφαλείας, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική ασφαλείας και δεν έχει και καμία σχέση με την πολιτική καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι ένα μέσο διαχείρισης της μετανάστευσης. Άλλωστε, η προέλευση του Γέροντα είναι εξής. εξή. Το σύστημα του Διβλίνου λέει ότι η πρώτη χώρα ε, και είναι αυτή η οποία υποδέχεται τον έτουντα άσυλο και είναι αυτή η οποία θα επεξεργαστεί την αίτησή του. Και πώς θα το ξέρουμε ότι είναι η πρώτη, φορά, πρώτη χώρα υποδοχής, ε, ζητώντας από κάθε άτομο το οποίο φτάνει να δώσει τα δαχτυλικά του αποτυπώματα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι από εκεί ε, μπήκε. Έτσι, αυτό το στόχο έχει το Eurodac. Αυτή τη στιγμή, και εδώ υπάρχει μια ανησυχία για την οποία ίσως να υπάρχει διάσταση απόψεων, ε, το θέμα δεν αφορά μόνο τα σύνορα, αλλά και τους ε, παράνομους που συλλαμβάνει η αστυνομία στις διάφορες χώρες. Ε, για ποιο σκοπό. Εάν οι αρχές Τη χώρα αυτή θεωρούσαν ότι είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει την ταυτότητά του και να δει αν έχουν ε, ε, μετακινηθεί από τη μία χώρα στην άλλη σε δευτερογενεί μετακίνησει, για να ξέρουμε και ποιο έχει την ευθύνη επαναπατρισμού εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν πλέον δικαίωμα να παραμείνουν σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Ε, η πιο απτή απόδειξη ότι το Eurodac δεν είναι μέσο ασφαλείας είναι γιατί δεν συνδέεται με το SIS που είναι το ε, κατεξοχήν ε, ε, ε, σύστημα ασφαλείας. Αυτό είναι το σύστημα, το SIS, μέσω αυτού τα κράτη-μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία σε εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι θα πρέπει ε, να τύχουν ειδική μεταχείρισης όταν εισέρχεται κάποιο στα σύνορα. Επιμένω σε αυτό διότι τίνουμε να το βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο και δεν θα ασχοληθούμε ίσως τόσο πολύ από τις συνθήκες ε, ε, εγγυήσεων εάν ε, οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν συστηματική πρόσβαση στη βάση δεδομένων. θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία στο πρόβλημα των 15 ημερών. Νομίζω ότι η πρόταση που έκανα είναι μια λογική λύση. Εξηγώ λίγο καλύτερα κύριε Πρόεδρε. Στο σύστημα Eurodac πρέπει να συμπεριληφθεί οτιδήποτε ε, εάν έχουμε ξεπεράσει την ημερομηνία ε, που προβλέπεται να παραμείνουν. Παραδείγματο χάρη, μία ομάδα φοιτητών που ε, έχασαν το αεροπλάνο του. αυτά δεν θα τα συμπεριλάβουμε στο σύστημα Eurodac. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν έρθει μόνιμα αυτοί που δεν έχουν ξεπεράσει από δεκα, κατά 15 μέρες την ημερομηνία που προβλέπεται να παραμείνουν δεν είναι απαραίτητο να φαίνονται όλοι στο σύστημα Eurodac. Εξαρτάται από την περίπτωση. Τώρα, αυτό που είπε η κυρία Χολμάχερ για τον αριθμό των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ε, λαμβάνω υπόψη με αυτό που είπατε για τα τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί? Γιατί η πιο πρόσφατη έκθεση των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βασίζεται και σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, το σύστημα εισόδου-εξόδου, λέει ότι με τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα έχουμε αρκετά στοιχεία και το πρόσωπο. Τα δέκα δακτυλικά αποτυπώματα είναι αυτά τα οποία προβλεπόταν από την ίδρυση του, σύσταση του συστήματος. Το πρόβλημα δεν είναι να περιοριστούμε στα τέσσερα. Το πρόβλημά μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό κανόνα γιατί την επαύριο θα συνδέονται τα συστήματα, θα συστέεται το Eurodac με το σύστημα εισόδου-εξόδου, τουλάχιστον να υπάρχει ένα κοινό κανόνα. Δεν είναι λογικό να λέμε ότι στο Eurodac πρέπει να έχουμε δέκα δαχτυλικά υποτυπώματα όταν δεν χρειάζεστε καν 10 αν δεν συμφωνούμε από αυτό, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής να μας πούνε τι λύση προτιμούν. Προσωπικά θεωρώ ότι τα τέσσερα αρκούν. Αυτά κύριε Πρόεδρε ε, ήθελα να πω. Α, α. Και η τελευταία ερώτηση του κυρίου Ντενανό για τα υποχρεωτικά δαχτυλικά αποτυπώματα. Θα είμαι λίγο προκλητικός τώρα εδώ κύριε Ντενανό. Αλλά αν το αφήσουμε αυτό στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών για το κατά πόσον θα πρέπει να πάρουμε τα δακτυλικατικά αποτυπώματα, ε, καλύτερο δεν θα ήταν να έχουμε μία ε, διάταξη ευρωπαϊκό επίπεδο παρά να αποφασίζει ο κύριος Ορμπάν και ο κ. Ορμπάν και όποιο έρθει στη συνέχεια. Αν σκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα για τέτοια προβλήματα, υπάρχουν κάποιε περιπτώσει ε, οι οποίε είναι τελείω διαφορετικέ. Στι δημοκρατικέ χώρε, στι πραγματικά δημοκρατικέ χώρε όπου υπάρχει μεγάλη προστασία και συστηματική, ναι. Αλλά κάποια χώρα που εκτρέπεται λίγο από τη δημοκρατική οδό, ίσω πρέπει να ε, τη ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω και κάτι ακόμα. Το ξέχασα. Ερώτηση του κυρίου Ντενανό πάλι που θεωρεί ότι δεν θα πρέπει ε, τα άτομα τα οποία ζητούν ε, διεθνή προστασία ε, και έχουν μετεκατασταθεί δεν θα πρέπει παρατήτως να διαβάζονται στο σύστημα Eurodac. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο σας παραπέμπω για τη μετεγκατάσταση, ζητά ανοιχτά να συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα Eurodac ιδιαίτερος για τους ελέγχους για τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι άκουσε προσεκτικά τις απαντήσεις σας ο κ. Στονανό. Έχει κάτι να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Όχι. Α, ναι, κάτι έχουμε. Λέγομαι Στρέλα. Ανήκω στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. θετική η γνωμοδότησή σας, οι τροπολογίες επίσης είναι σταθμισμένες. Το Συμβούλιο και δεν αμφιβάλλω ότι και η Επιτροπή θα τα εξετάσει προσεκτικά όταν ξεκινήσει ο τριγωνικός διάλογος. Κάποια σχόλια παρακαλώ για τον αριθμό των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το Eurodac απαιτεί όπως ξέρετε το σύνολο των αποτυπωμάτων και αυτό δικαιολογείται από τον στόχο τον οποίο έχει να πετύχει την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Ο κίνδυνος λανθασμένου εντοπισμού που θα μπορούσε να μετεφερθεί ε, για κάποιον σε μια άλλη χώρα ε, είναι υπερβολικός κίνδυνος και θα δημιουργήσει νομικά προβλήματα. Είναι θέμα λοιπόν αξιολόγησης κινδύνου και ακρίβειας. Στην περίπτωση του Eurodac, ακόμα και τη στιγμή που θα έχουμε αλφανιουμέρικ δεδομένα, μιας και αυτού του είδους τα δεδομένα ε, δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα αξιόπιστα, και απαιτείται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια και η ακρίβεια αυτή παρέχεται από τα 10 δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί ιστορικά χρησιμοποιεί το Eurodac τα 10 δάχτυλα. Γιατί όταν σχεδιάστηκε ήταν η πρακτική σε πολλά κράτη-μέλη στις δυνάμεις ε, εφαρμογής της τάξης, τήρησης της τάξης να παίρνουν τα αποτυπώματα και των δύο χεριών, των μετακινουμένων. Τα εθνικά συστήματα εργάζονται πάντα σε βάση 10 αποτυπωμάτων. Να πω επίσης ότι η Eurodac είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί διαλειτουργικά, μειώνοντας τον αριθμό των αποτυπωμάτων, μπορεί να βοηθήσουμε ίσως την διαλειτουργικότητα με άλλα σύστηματα, αλλά νομίζω ότι υπονομεύουμε ε, την συγκρισιμότητα στο εσωτερικό του Eurodac. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, μένουμε εκεί κύριε Σιγητά. Οι τροπολογίες λοιπόν θα κατατεθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, τις 5 το απόγευμα. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει στις 6 Μαρτίου και η ψηφοφορία στη Λίμπε θα γίνει στις 30 Μαρτίου. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση του κυρίου Ντεπρέ, τον αριθμό 16, για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την κατάθεση ή μάλλον για την εξέταση μιας αίτηση που έχει κατατεθεί για διεθνή προστασία από πλευράς ενός απάτριδος ή ε, προσώπου πολίτη τρίτης χώρας. Είναι ένα θέμα λίγο πιο περίπλοκο αυτό από ότι το προηγούμενο. Γνωρίζετε πως έχει κατάσταση. Ε, βιώνουμε ακόμα το Δουβλίνο 1 που καθιστά την πρώτη χώρα που υποδέχεται τον πρόσφυγα η υπεύθυνη χώρα για την αντιμετώπιση της αίτηση και των συνεπειών αυτής. Το Δουβλίνο είναι άνισο σε σχέση με τις χώρες που υπάρχουν. Ξέρετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα Ξέρετε ότι έχουν τεράστιους αριθμούς ετούντων άσυλο. Η Επιτροπή καθορίζει έναν μηχανισμό διορθωτικό, δηλαδή έναν μηχανισμό ο οποίος θα κατανείμει αυτούς που ζητούν άσυλο μέσω ενός ε, τύπου, αν θέλετε, αλληλεγγύης ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Ένας διορθωτικός αλληλέγγυος μηχανισμός. Καταρχάς ο μηχανισμός αυτός τίθεται σε λειτουργία αν θέλετε με βάση συγκεκριμένους κανόνες και αυτή τη στιγμή ένα κράτος μέλος και σπάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας φτάσει το 150% της δυνατότητας υποδοχής η οποία του αναλογεί. Δηλαδή αν είχε 100.000 θα πρέπει να φτάσει στους 150.000 για να λειτουργήσει αυτός ο διορθωτικός μηχανισμός. Δηλαδή αφήνουμε στις πιο εκτεθειμένες χώρες 50% επιπλέον της δυνατότητας υποδοχής που τους αναγνωρίζουμε, πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός διόρθωσης. Εγώ θεωρώ και σας το εξηγώ ότι ο κανόνας αυτός δεν είναι διόλου σοφός, γιατί οι χώρες που έχουν την πιο βαριά ευθύνη θα συνεχίσουν να έχουν την πιο βαριά ευθύνη, την οποία ο ίδιος ο μηχανισμός καθορίζει. Συνεπώς λοιπόν ο διορθωτικός μηχανισμός κατανοής, κατανομής να ξεκινάει στο 100% και όχι στο 150%. Αυτή τη στιγμή κατέβουν στο 90% και παίξει ο μηχανισμός αυτός, τότε θα ξεκινήσουν πάλι την υποδοχή προσφύγων. Λοιπόν, γιατί κάνω την πρόταση αυτή. Γιατί αν πάρετε τον κανόνα του 100 και όχι τον κανόνα του 150, σαν σημείο εκκίνησης της λειτουργίας του μηχανισμού. Ο μηχανισμός θα λειτουργήσει νωρίτερα και αυτό θα έχει πιο σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες. Δεύτερη αλλαγή. Η Επιτροπή προβλέπει κάθε φορά που κάποιος που ζητά άσυλο ή που αιτείται διεθνούς προστασίας επαναγκαθίσταται κάπου, και μεταφέρεται σε μια άλλη χώρα στα πλαίσια του μηχανισμού αυτού, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα δώσει 500 ευρώ για κάθε άτομο στην χώρα η οποία θα μεταφέρει τον συγκεκριμένο πολίτη. Αν η Ελλάδα στείλει κάποιον στην Πολωνία σαν παράδειγμα ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία, η Ελλάδα θα πάρει 500 ευρώ. Περίεργο μου φαίνεται αυτό. Για δύο λόγους. Πρώτον, θα μπορούσαμε ακριβώς να δώσουμε την δυνατότητα κάποιου χρηματικού κέρδους, ε, γιατί αυτός θα είναι που θα πληρώσει τη μεταφορά. Δεν θα πρέπει να είναι σώνη και καλά εις βάρος ε, της χώρας που υποδέχεται. Γιατί 500 ευρώ μου είπαν ότι δεν υπάρχει κριτήριο, είναι μια εφάπαξ πληρωμή, καταποκοπήν συγγνώμη πληρωμή. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό να το κάνει κανείς, γιατί έχουμε κάθε συμφέρον. Λέμε ότι το καταποκοπή να μην είναι 500, να είναι 300 ή 200, γιατί η βοήθεια προς τις χώρες αυτές γίνεται με άλλους μηχανισμούς, όπως με τις έκτακτες επιδοτήσεις τις οποίες γνωρίζαμε τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή η πρόταση αυτή γιατί επαναλαμβάνω υπάρχει βοήθεια πιο λειτουργική και άλλης μορφής υπέρ χωρών όπως η Ελλάδα και της Ιταλίας επίσης. Τρίτον, το πιο αν θέλετε σημαντικό για μένα που θα προκαλέσει συζητήσεις. Η Επιτροπή μας λέει ότι όταν ένα κράτος μέλος αρνείται να πάρει μέρος στο διορθωτικό μηχανισμό θα επιβληθεί σε μια ποσόστοση ας πούμε 2.000 ε, και υποτίθεται ότι πρέπει να πάρει 100, ε, η Επιτροπή λέει πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο. 250.000 ευρώ κατά κεφαλήν. Αν μπούμε στο σύστημα φυσικά των, ε, των προστήμων, το κράτος πληρώνει. Ε, το κράτος σας υποθέσουμε ότι δεν πληρώνω, διότι η κατάστασή μου δεν μου το επιτρέπει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς κολυσιεργίας και δικαστικούς, λέγοντας ότι το πρόστιμο το οποίο ε, μου ζητείτε να πληρώσω δεν είναι ε, τεκμηριωμένο. Αντί λοιπόν για ένα τέτοιο σύστημα, εγώ θα προτιμούσα ένα σύστημα ας πούμε προπληρωμής, δηλαδή στα διάφορα των διαφόρων ταμείων όπως το Ταμείο Συνοχής και τα λοιπά, θα αφαιρείτε ένα ποσό για τις χώρες που αρνούνται να πάρουν μέρος στο μηχανισμό αλληλεγγύης. Γιατί όταν έχετε έναν μηχανισμό αλληλεγγύης και τιμωρηθείτε, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν είχατε θεωρητικά την επιλογή εφόσον είναι υποχρεωτικός. Οπότε η κύρωση θα πρέπει να είναι άμεση και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει η συνέπεια να είναι η αφαίρεση ας πούμε του 10% των ποσών του Ταμείου Συνοχής που έχετε ανάγκη. Ξέρω ότι η επιλογή αυτή την θέτω προσυζήτηση Ίσως να μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός πιο διαφθρωμένος και πιο αποδεκτός, αλλά ε, μια αυτόματη παρακράτηση, αν θέλετε, ενός ποσοστού είναι θα έλεγα πιο αποτελεσματική από μια στρατηγική ε, προστίμου. Γιατί το πρόστιμο δεν είναι εγγυημένο ότι θα πληρωθεί. Ενώ η προπληρωμή, η παρακράτηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει κεντρικά. Και οι χώρες φυσικά αυτές θα βοηθήσουν τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στον ε, μηχανισμό αυτό κατανομής. Μιλάμε για μια πραγματική ε, αμοιβεοποίηση. Δυστυχώς πρέπει να σας ε, εγκαταλείψω, λέει ο Πρόεδρος, λυπάμαι γιατί η συζήτηση έχει νόημα και θα έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό να ζητήσω και πάλι από τον κύριο Άνσουορθ να αναλάβει πάλι την Προεδρία. Ζητώ συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να παραμείνω άλλο. να ευχαριστήσω τον κύριο εισηγητή. Πράγματι η πρόταση που κάνατε είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα προς αναζήτηση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Τρεις ομιλητές έχω στον κατάλογο. Η κυρία Σολάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Σδεχόφσκι είναι είναι σκιώδης ηγητής μας και μου ζήτησε να παρέμβω εξ του. Ο Σκιώδης της ευχαριστεί τον κύριο Ντεπρέ για τη δουλειά του, αλλά δεν ε, συμφωνεί με τις ε, τροποποίησεις που προτείνει. Με εξαίρεση τη διαλειτουργικότητα. Ο κύριος Δεκόφσκι απορρίπτει την ιδέα χρηματοδότησης ε, του αποθεματικού του Δουβλίνου με 10% των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν τηρεί τις υποχρώσεις του. Ο μηχανισμός αυτός δεν θα έπρεπε να αφορά την πολιτική συνεχής και καμία άλλη πολιτική. Ο κύριος Δεχόφσκι θεωρεί ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού όταν φτάνουμε στο 100% ε, ίσως ε, θα μπορούσε να το συζητήσει και να βρούμε κάποιο συμβιβασμό. Γιατί προβλέπεται από εκεί και πέρα αναστολή του μηχανισμού όταν φτάνουμε στο 90% των δυνατοτήτων. Κατά τον άποψή του το, όριο θα πρέπει να είναι το 100%. Τρίτο σημείο. Κύριος Δεκόφσκι. διαφωνεί ε, στη μείωση των δαπανών από 500 σε 300 ευρώ για κάθε πρόσφυγα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χόλμαϊερ. Το Δουβλίνο θα μας απασχολήσει σίγουρα και τα ακόμα. Και θα πρέπει να βρούμε μια λύση με τα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη συμφωνούν πιο πολύ παρά ποτέ και είμαι αρκετά σαρκαστική γιατί εδώ το συζητάμε 15 χρόνια και εγώ 7 χρόνια προσωπικά για το Δουβλίνο και ω τώρα τα κράτη-μέλη έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε λύση παρά το γεγονός ότι βλέπουν ότι μας οδηγεί στην καταστροφή αυτό το θέμα. Και μάλιστα αυτό διακυβεύει και τις κοινέ αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί οι επιδράσεις, οι επιπτώσεις ε, του να μην επιληθεί το Δουβλίνο και το μεταναστευτικό ζήτημα σημαίνει ότι θα έχουν όλο και πιο πολλού καυγάτε μεταξύ του και αντιπαραθέσει τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι διαφέρει κάπως η άποψή μου από αυτή τους κοιόδους μα. Πώς καταλήγουμε στα 300 ευρώ. Και νομίζω ότι στο ιστορικό της Ευρώπης δεν ε, είναι τόσο ακριβά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τόσο υψηλό το κόστος για την αλληλεπρέωση των αιτήσεων των προσφύγων. Και θα πρέπει λοιπόν να συνομιλούμε επί μιας αντικειμενικής βάσης. Το θέμα του παθηματικού για το Δουβλίνο μου προκαλεί κάποιες απορίες από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών έχουμε μία προσέγγιση η οποία δεν είναι συγκεκριμένη μόνο για τα ταμεία συνοχή, αλλά τι λέει, ότι ένα κράτο μέλο, αν δεν πληρώσει τα πρόστιμά του, πολύ απλά αυτά αφαιρούνται από τα ποσά τα οποία θα λάμβανε το κράτο μέλο. Και αναρωτιέμαι, αυτό αναφέρεται μόνο στο Ταμείο Συνοχή, γιατί υπάρχουν ταμεία, χώρε που δεν χρησιμοποιούν τα Ταμεία Συνοχή. Ποιο είναι ο κανονικό μηχανισμό λοιπόν που υπάρχει στο... Μήπως θα μπορούσε να, συ... εφαρμοστεί η αρχή που εφαρμόζεται έτσι και αλλιώς στον έλεγχο προϋπολογισμών και για το Δουβλίνο. Και αυτό όμως να μην πλήξει μόνο τις χώρες ε, που λαμβάνουν κονδύλια από ταμεία συνοχής, γιατί υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες δεν λαμβάνουν διαφορετικά ταμεία συνοχής, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι επικοδομητικές. Και έτσι λοιπόν, ε, αν κάποιος ε, δεν έχει πληρώσει το πρόστιμό του, αυτό ενδεχομένω να μπορεί να αφαιρεθεί από τις επιδοτήσεις στη γεωργία ή οποιονδήποτε άλλο τομέα. Και έτσι θα μπορούσε να αφαιρέσει η Ένωση τα ποσά αυτά. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι θα λειτουργούσε καλά και θα μιλήσουμε για την Μιλάμε για ποσά 52.000. Να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς καταλήγει στο πόσο αυτό. Στη Βαβαρία θεωρώ ότι δεν θα έφτανε το 52.000. Και αν σκεφτώ το τι δυνατότητε έχουν κάποιες χώρες, θεωρούμε ότι τα 250.000 είναι υπερβολικά ψηλό ποσό. Πώς καταλήγεται λοιπόν, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ποσό αυτό. Και θα, προσπα... πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία συγκεκριμένη τέτοια μέθοδο στις ε, αναλύσεις μας. Ε, υπάρχουν υποχρεώσεις λοιπόν, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν. Και αν είναι απονομικής άποψη τα πράγματα έτσι, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για κάποιο πρόστιμο, το οποίο είτε θα καταβάρεται στην Ένωση ή θα αφαιρείται από κάπου αλλού. Κανονικός και φυσιολογικός μηχανισμός. Αλλά δεν είναι μόνο για τις ε, χώρες συνοχής ε, και για άλλες συγκεκριμένες χώρες. Επίσης, να υπογραμμίζω το εξή. Δεν είναι μόνο οι χώρες στην πρώτη γραμμή αυτές που πλήττονται. Η Γερμανία έχει τους πιο πολλούς πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είμαστε ούτε στη Μεσόγειο, ούτε στην πρώτη γραμμή. Και παρόλα αυτά έχουμε υποδεχτεί τους πιο πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες. Άρα το όλο σύστημα θα πρέπει να το εξετάσουμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά ε, την πρώτη γραμμή. Και το Βέλγιο έχει πάρα πολλούς ε, μετανάστες. Μην το ξεχνάμε όχι όλοι καταχωρισμένοι. Θα πρέπει λοιπόν το σύνολο του μηχανισμού να λειτουργεί. Για το λόγο λοιπόν αυτό θεωρώ ότι είναι καλό το γεγονό ότι ξεκινάει αυτή τη συζήτηση ω ραντεπρέ για να κάτσουμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν μόνο ένα κομμάτι των κρατών μελών να αναλαμβάνει τις υποχρέωσει υποχρεώσεις αυτές οι άλλοι να κάνουν την πάπια και η τρίτη ομάδα να κάνει ό,τι θεωρεί αυτή σωστό και να προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις. Είχε γίνει και η εξή πρόταση, ότι αν ένα κράτος μέλος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και πάνω από το 100% αρχίζει να συζητάει θέματα ανακατονομής, αυτό θα μπορούσε να με βρει σύμφωνη, θα μπορούσα να κατανοήσω και κάτι άλλο που θεωρώ ότι είναι θετικό, κάτι που είναι στο τέλος τέλος. Για τον διευθυντικό μηχανισμό, αν ένα κράτος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και γίνεται ανακατανομή χωρίς να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, είναι κάτι το οποίο θα θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη της προς τα άλλη κράτη-μέλη. Και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Ευχαριστώ, Μόνικα. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική στιγμή ε, ο καλύτερος τρόπος να έχουμε περισσότερους αντιευρωπαίους από ό,τι σήμερα. Η χώρα μου αναφέρθηκε αρκετές φορές και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ειδικά του μηχανισμού αυτού. Ε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καταρχάς, διότι ήδη με τις 250.000 έχουν εκτοξευθεί τα πράγματα ε, στη δημόσια συζήτηση. Ο κόσμος είναι οργισμένος ε, γιατί πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Και δεύτερον, ο σαφή σύνδεσμο με την πολιτική συνοχή, που στην πραγματικότητα είναι η άλλη πλευρά τη ενιαία αγορά και είναι οι μακροοικονομικέ μεταφορέ. Δεν είναι τα χρήματα τα οποία καταβάλει κάποιο για να σου τα πάρει, γιατί δεν σου τα έχει δώσει. Είναι μια μεταφορά που έχει σχέση με την ενιαία αγορά. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, ε, ε, βάσει του σημερινού κανονισμού δεν είναι νόμιμο Εκτό μικροφώνου τα σχόλια τη κυρία Χολμάλια. Με τα υπόλοιπα όμω, ναι. Αν έχουμε τα εθνικά χαρτοφυλάκια, υπάρχουν οι δεσμεύσει και βάσει και των δεσμεύσεων έχουν υπογραφεί και συμβάσει ε, και υπάρχουν επενδύσει εν εξελίξη, αυτή είναι δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ουσιαστικά ε, το θέμα δεν είναι να ξαναδούμε όλο το μηχανισμό. το θέμα είναι να δούμε σε ποιο σημείο έρχεται η υποχρέωση των κρατών μελών και η συμφωνία όλων των κρατών μελών για μια κοινή υποχρέωση που οδηγεί και σε συνέπειες. Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αφορά το Ταμείο Συνοχής ή Κονδύλια Συνοχής, γιατί το, αν είναι Κονδύλια Συνοχής αφορά όλες τις χώρες, αν είναι Ταμείο Συνοχής αφορά την κάθε χώρα. Νομίζω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί αυτό, γιατί αλλάζει η κατάσταση. Παραδείγματο χάρη, στη χώρα μου. Έχουμε τα πρώτα ε, στοιχεία για παράνομους μετανάστες που έρχονται από την Ουκρανία. Θέλουν να πάνε στη Γερμανία βεβαίως και κανονικά βάσει Δουβλίνου πρέπει να τους σταματάμε εμείς στην Πολωνία. Δημιουργείται λοιπόν μια εντελώ νέα κατάσταση. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα. Το πρόβλημα της αλληλεγγύης επήγει, αλλά το να πρέπει να πληρώσουν τα κράτη-μέλη ή να τους περικόψουμε χρήματα είναι ένα από τα πιο λογικά στοιχεία τα οποία θα έχουμε σε επόμενους μήνες. Δεν νομίζω ότι βέβαια αυτό είναι το τέλος της συζήτησης, μάλλον στην αρχή είμαστε, αλλά ήδη αυτές οι 250.000 ε, οδήγησαν σε πολύ μεγάλη απογοήτευση στη δημόσια συζήτηση και το επόμενο ερώτημα είναι το Ταμείο Συνοχή. Νομίζω ότι όλα αυτά θα έρθουν με τη συζήτηση για το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν έχω καμία αμφιβολία περί τούτου. Αλλά ε, ίσω θα έπρεπε να ε, έχουμε μια ανακατανομή στον προπολογισμό για να είναι πιο ευέλικτο. Βάσει του σημερινού προπολογισμού, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά κυρίω στο Συμβούλιο να περάσουν όλα αυτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκαρδιαθαμπάλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα, γιατί ε, λιγοστεύουμε και πάμε. Σήμερα το απόγευμα ε, αυτά τα θέματα τα οποία είναι τελικά θέματα πολιτικών ελευθεριών περισσότερο παρά προπολογισμό, μάθαμε πολλά για το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα το πώ μεταφράζονται όλα αυτά σε προπολογισμό είναι πολύ ωριακά. Εμεί κάνουμε μια πιο γενική συζήτηση νομίζω ε, για αυτά τα οποία συζητούνται και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών παρά ε, για τη συνέπειε στον προπολογισμό. Παρά το γεγονό ότι ανάλογα με τι αποφάσει που θα λάβουμε θα υπάρξουν και συνέπειε στον προπολογισμό. Εμεί από πλευρά μα να πούμε ότι συμφωνούμε ε, να... περάσουμε στο 100% από το 150% για το, ε, ε, την ενεργοποίηση της διόρθωσης, ε, την εξήγηση μας την έδωσε ο κύριος Ντεπρέ, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Ε, δεν θέλουμε να πάμε στο 90%, ίσως ακόμα και στο 80% για να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο σε χώρες οι οποίες θα έχουν συνεχώς, θα βρίσκονται εντός ή εκτός του συστήματος. Και όσον αφορά την τελευταία συζήτηση, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα για το τι πρέπει να κάνει όταν ένα κράτος μέλος ε, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να του επιβληθούν κυρώσεις. Πρώτα-πρώτα μου φαίνεται εντυπωσιακό να συζητάμε κατά πόσον ένα κράτος μέλος μπορεί ή όχι να τηρήσει ένα νόμο ο οποίος θα εγκριθεί από εμά. Και από εκεί και πέρα το να μην υπάρχουν κυρώσεις ε, ε, είναι αδιανόητο. Γι' αυτό και κατανοώ αυτό που λέει και ο κύριος ε, Ντεπρέ, που λέει ότι υπάρχει πολύ πιο εύκολος τρόπος να υπάρχει μία προειδοποίηση, να είναι κάτι πιο αυτόματο από ένα πρόστιμο. Ε, από ό,τι κατάλαβα θα είναι από το Ταμείο της Συνοχής εγώ, που σημαίνει ότι θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα κράτη-μέλη, ε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ λογικό. περισσότερο μάλλον στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών από ότι εδώ θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς μπορεί να επιβληθεί κύρωση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές οι κυρώσεις. Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις και επομένως και η νομιμότητα ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν σε ένα λεπτό, αλλά πριν θα ήθελα να πω στον εισηγητή, καταρχάς ευχαριστώ. Όπως είπε και η Αίντερ, είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και χαίρομαι και κρίμα που δεν έχουμε και τόσους πολλούς συναδέλφους εδώ, αλλά όπως είπε και ο εισηγητής, είναι κοινό το πρόβλημα, όλα τα κράτη-μέλη το έχουν και Το ένα θέμα είναι το πόσο εκτεθειμένα είναι τα κράτη-μέλη στο θέμα και διαφορά στην έκθεση είναι αυτό το οποίο ε, ε, αλλάζει τα πράγματα και τα κονδύλια τα οποία έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικά, κυρίως για κράτη που εξορισμού δεν έχουν τόσα χρήματα. Σίγουρα είναι θέμα αλληλεγγύης, αλλά όπως και αρκετοί συνάδελφοι είπαν, είναι και η ισότιμη μεταχείριση ε, για τις χώρες αυτές και αντίστοιχη αλληλεγγύη. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει να μας πει. Εγώ... Αντικαθιστώ μόνο τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνα για το θέμα αυτό. Είναι άλλο επιτροπή. Η γνώμη μου εδώ δύσκολα εκφράζεται για οποιαδήποτε πρόστιμα και κυρώσεις, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα. Φτιάχνουμε ένα σπίτι και ξεκινάμε από την καμινάδα. Δεν έχουμε ακόμα ρίξει τα θεμέλια. Ούτε ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν. Δεν ξέρουμε ποιος θα αποφασίσει και τι. Η δική μου χώρα, για παράδειγμα, υποδέχεται πολλούς από την Ουκρανία, αλλά τώρα δεν φαίνεται να είναι της μόδας οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Πιο πολύ μιλάμε για τους ε, Σύριους κτλ. Δύσκολα λοιπόν μπορώ να εκφράσω την ε, άποψή μου για το τι θα γίνει και πώς θα τιμωρηθούν τα κρατημέλη που δεν θα υποδεχτούν τους πρόσφυγες που του αναλογούν και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρουμε ποιος ε, θα είναι. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη γιατί κοιτούσα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν κατάλαβα ότι ήσασταν και εσείς εκεί ως αναπληρωτής στην Επιτροπή ε, Προπολογισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Να σχολιάσει. Θα σα ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Είμαι επικεφαλή στην Γενική Διεύθυνση Μπάτζ. Θα σχολιάσω το θέμα της μετάβασης από το τέλος αλληλεγγύης σε ένα 10% ενδεχομένως. Και μετά θα μας ε, πει και δύο-τρία πράγματα ως συναδελφός από την Δυτικό. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε να σας πούμε ότι έχουμε και κάποια ερωτηματικά, τα ανέφεραν και κάποιοι άλλοι και κάποιοι βουλευτές για το είδος των, ε, της χρηματοδότησης που συζητάμε. Γιατί δεν καλύπτονται όλα τα κρατημέλη, δεν λαμβάνουν όλα τα κρατημέλη ταμεία συνοχής. Μιλάμε και για άλλα περιβαλλοντικά ταμεία λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Κατά δεύτερον, θα δημιουργηθεί σύνδεσμος μεταξύ δύο διαφορετικών πολιτικών που δεν ήταν απαραίτητα η αρχική πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενδεχομένως λοιπόν να πρέπει να τσεκάρουμε και τη νομική εφικτότητα ενό τέτοιου μηχανισμού. Και τέλο, θα δημιουργηθούν και κάποια ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική διαδικασία, γιατί ενδεχομένω αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβερθούν κάποιε κονδύλια σε διαφορετικά κεφάλαια και αυτό ενδεχομένω να είναι περίεργο. Είμαστε μάλλον διστακτικοί λοιπόν για αυτή την πρόταση. Και έχουμε και κάποια άλλα σχόλια για κάποιες άλλες προτάσεις. Σας ευχαριστώ για να τάμλε από την ε, Γενική την Home Affairs ε, για τις 250.000. Ε, ρωτήσατε πώς το υπολόγισε αυτό το ποσό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι δεν έγινε αμίγως επιστημονική ε, μελέτη και υπολογισμό, αλλά έχουμε δύο στοιχεία που μα οδήγησαν στο ποσό αυτό. Καταρχά, υπολογίστηκε το κόστο το οποίο θα ε, επιβαλλόταν στο κράτο μέλο για την υποδοχή ενό ε, μεταναστή πρόσφυγα για κάποια χρόνια. Και κατά δεύτερον, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη στον ερωτικό μηχανισμό. Είναι ένα αποτρεπτικό παράγοντα και γι' αυτό λοιπόν καταλήξαμε στα 250.000 χιλιάρικα το θέμα του κόστους μεταφοράς, 500 ή 300 ευρώ ως πόσο καταποκοπεί. Ναι, επιλέξαμε τα 500 ευρώ γιατί αυτό είχε αποφασιστεί από την απόφαση μετακατάστασης για την Ελλάδα και την ε, Ιταλία και πάλι δεν υπήρχε κάποια επιστημονική βάση. Θα μπορούσαμε να το χαμηλώσουμε το πόσο αυτό, αλλά καλά θα ήταν να υπάρχουν και κάποια στοιχεία για το πραγματικό κόστος. Τώρα να πούμε δύο λόγια για το δανειοδοτικό μηχανισμό, για το 100-150% ή μάλλον μια διευκρίνηση καλύτερα. Αυτό το 100% δεν αφορά την ε, ικανότητα υποδοχή του κράτου μέλους, αφορά την, ε, το δίκαιο τμήμα και μερίδιο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί είναι σημαντικό σε όλο το σύστημα να καταλάβουμε τι λέμε. Α υποθέσουμε. Α, όχι, καταλαβαίνετε. Okay. Δεν σημαίνει ότι έχει εξαντληθεί 100% η δυνατότητα υποδοχή ε, του κράτους μέλους. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι το ποσό που του αναλογεί, το, ο όγκος που του αναλογεί και μπορεί να είναι χαμηλό ως αριθμητικό στοιχείο. Αν πάμε στο 90% ή στο 80% αυτό τι θα σημαίνει ότι το κράτος μέλος θα έκανε λιγότερα από αυτά που του αναλογούν από το δίκαιο μερίδιο που του αναλογεί και γι' αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε και το 150% για την κινητοποίηση και την ε, ανακοπή και αναστολή του μηχανισμού. Τελευταίο θέμα για τη δυνατότητα αναστολής σε περίπτωση ανεπαρκών ελέγχων στα σύνορα. Είπαμε δύο τρίτα πλειοψηφία στο Συμβούλιο και η συνένεση του Κοινοβουλίου. Αυτό προβλέπεται. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και από πλευρά νομική εφικτότητα, γιατί πλέον υπάρχει ένα νούμερο κλάουζο σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε αυτέ στην συνθήκη. Και δεν βρήκαμε πουθενά να προβλέπεται δύο τρίτα πλειοψηφία. Αυτό από νομική αμυγό άποψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο, και τώρα το λόγο έχει ο εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το σύνολο των συναδέλφων που πήραν μέρος στη συζήτηση. Είχα πει στην αρχή ότι η συζήτηση αυτή είναι πιο δύσκολη. Θα ξεκινήσω λέγοντας προς τον Γιάνν και προς άλλους συναδέλφους ότι εμείς είμαστε το Κοινοβούλιο. Εγώ γνωρίζω τους δισταγμούς του Συμβουλίου, αλλά δεν θα το παίξουμε Συμβούλιο. Έτσι όπως έχει το, η κατάσταση προσπαθούμε να καθορίσουμε την θέση του Κοινοβουλίου. Ποια θα είναι η τελική θέση τώρα, αυτό θα φανεί Προσπαθώ να καθορίσω λοιπόν τη θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με την αρχική πρόταση. Όλα τα σημεία τα οποία τέθηκαν είναι υποσυζήτηση. Εγώ αν θέλετε να κάνουμε μια μεγάλη συνάντηση, να μιλήσουμε για 100%, 150%. Υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παντού. Για τα έξοδα μεταφοράς. Δεν υπάρχουν, δεν έχετε κριτήρια αντικειμενικά, ούτε και εγώ έχω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, μηχανισμοί βοήθειας προς τις χώρες πρώτης γραμμής. Ε, αυτό λύνει το θέμα. Είστε αυθαίρετοι εσείς, είμαι ε, και εγώ αυθαίρετος και το θέμα είναι να προσπαθήσει κανείς να είναι όσο αυθαίρετος, στο λιγότερο αυθαίρετος μπορεί να γίνει για να μην υπάρχει μεγάλο κόστος. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για τα ταμεία συνοχής. Τα ταμεία συνοχής λοιπόν. Το πρόβλημα είναι το εξής, επαναλαμβάνω. Ένας διορθωτικός μηχανισμός και ένας μηχώνας ελεγγύης, μηχανισμός ελεγγύης δεν είναι κάτι το εθελοντικό. Όλες οι χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και οι δικοί μου, συνεισφέρουν στην τροφοδοσία των ταμείων συνοχής. Υπάρχει ένα στοιχείο δηλαδή εδώ αλληλεγγύης. Εγώ δεν αρνούμαι ε, την ε, λογική της ε, οργάνωσης της αγοράς αυτής και της συνοχής. Υπάρχει λοιπόν ένα στοιχείο αλληλεγγύης στον τομέα της συνοχής. Όποιος δεν δέχεται την έννοια της αλληλεγγύης σε έναν τομέα, τότε υφίσταται τις συνέπειες σε έναν άλλο τομέα. Εγώ είπα 10%. Μπορείτε αν θέλετε να τα υπολογίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Να πούμε ότι θα αποσύρουμε επιστώσεις πληρωμής σε ένα ποσό το οποίο να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ανθρώπων που δεν έγιναν δεκτοί από μια χώρα πολλαπλωσιασμένο κατά 150.000 λέω τώρα. όπου ερχόμαστε σε έναν μηχανισμό ακριβώς ε, προστίμου, γιατί μια χώρα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει δικαίωμα να μην τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κινδυνεύει να ισχύσει για πάρα πολλά χρόνια. Αν η Μόνικα έχει μια καλύτερη λύση, την ε, δέχομαι την λύση αυτή. Δεν έχω αμφιβολίες, δεν έχω δισταγμούς, δεν έχω copyright. Εγώ θέλω έναν μηχανισμό σχετικά αποτελεσματικό. Και γι' αυτό είμαι ανοιχτός σε συζητήσεις και σε προτάσεις. Πάντως γνωρίζω ότι το θέμα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει ιδιαίτερο στην προσοχή της Επιτροπής ΙΤΡΕ που βασίζονται σε θέματα αρχών και όχι τόσο σε θέματα δημοσιονομικά. Οπότε σε επίπεδο αριθμών εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι στην τελευταία σας παρατήρηση που νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας ε, περισσότερη επιλογή και όχι οι κυρώσεις. Ε, τα κράτη-μέλη επιλέγουν να μη συμμετέχουν, ουσιαστικά επέλεξαν να πληρώσουν αυτό το ποσό, αντί να πούν ότι δεν συμμετέχετε, άρα θα σας τιμωρήσουν. Αυτό είναι απλώς η απόψή μου βεβαίως. Να υπενθυμίσω στους αδέλφους λίγο το χρονοδιάγραμμα, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 15 Φεβρουαρίου, 5 η ώρα. ψηφοφορία 6 Μαρτίου στην Επιτροπή μας και στην επί της αρμόδια Επιτροπή στη ΛΥΜΠΕ ε, προσεχώς. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή και περνάμε στο σημείο 20 στην ημερήσα διάταξη τα διάφορα. Δεν βλέπω κάποιον να ζητάει κάτι. Επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα 6 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Θέλετε κάτι? Ε, απλώς με αποχαιρετάει, κύριε Δεπρέ. Πέρα συνεδρίαση.